αυτό γιατί η κατάσταση στην ε, Ιταλία, Σουηδία ή Πολωνία ε, σημαίνει ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ε, αλλού υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείε, αλλού δημόσιες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ακούσουμε την φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν γίνει αυτό λοιπόν θα είναι καλύτερος και ο κανονισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγο τώρα έχει ο κύριος Μαριάς το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτή την προοπτική και όχι βέβαια να αποτελεί εμπόρευμα και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ε, επιχειρηματικούς ομίλους. Και στη βάση αυτή θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο της επαναχρησιμοποίησης των υδάτινων πόρων διότι ε, υπάρχει τεράστιος περιορισμός στους υδάτινους πόρους έχουμε και την κλιματική αλλαγή που επιτείνει το πρόβλημα κατά την έννοια αυτή πρέπει να δούμε πώς θα επαναχρησιμοποιήσουμε ε, τα ύδατα πρέπει να μπουν σε μια λογική τέτοια που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος στην στήριξη της ε, δημόσιας υγείας. φυσικά η επαναχρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων σημαίνει υποδομές σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν και τα αντίστοιχα κονδύλια για να μπορέσει να υπάρξει η λειτουργία αυτή και κυρίως σε μια κατεύθυνση τέτοια που να στηρίξει την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος ένας ομιλητής, Νέκοφ. Παρακαλώ. Πράγματι, το νερό δεν είναι ένα κοινό αγαθό, σαν πολλά άλλα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο και η αστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα οι πρωτεύουσε ε, δημιουργούν σημαντικές εντάσεις και πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να τις μειώσουμε αυτές τις πιέσεις και μία λύση θα ήταν η ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης των λιμάτων. Ο γεωργικός τομέας είναι παράδειγμα Θα ήταν πολύ σημαντικό όμως να αποφύγουμε τη μόλυνση των εδαφών μέσω του νερού, ιδιαίτερα με μικροπλαστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νέκοφ. Ε, α, έχουμε και τη στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω, όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένω ότι η ένταξη το Ρωμά είναι υποχρέωσή μα και πρέπει να ξεπεράσουμε τη λογική ότι τόσα εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, ιδίω σε συγκεκριμένε περιοχέ τη Ιταλία, στην Ήπεθρο α πούμε, αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Είναι ένα πρόβλημα που εμένει. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και πολλέ φορέ δεν λαμβάνεται καν υπόψη στο σύνολό του και σε όλο σε όλο το μέγεθο. Τα δικαιώματα που υπάρχουν και τα κονδύλια που προσφέρονται για την αντιμετώπιση τέτοιων προγραμμάτων, τέτοιων προβλημάτων, είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Προτεραιότητα λοιπόν πρέπει να δοθεί σε αυτή τη στιγμή σε όποιον δεν έχει δουλειά και ψάχνει και να τους δώσουμε την ευκαιρία να τη βρουν. Kiitokset edustaja Olkaa hyvä. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για την στρατηγική ένταξη ε, των Ρωμά. Πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και συμφωνώ και με τους κύριους στόχους ε, της στρατηγικής, ε, όπως απασχόληση, στέγαση, υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέθεσε κι άλλον έναν στόχο, την διακριτική μεταχείριση. Ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει η Πρόεδρος, ε, δεν ακούγονται τα φιλανδικά. Να τα ξαναπώ. Α, τώρα ακούγονται, εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω τα μόλις ε, τα όσα ανέφερα μόλι τώρα. Υποστήριξα την έκθεση αυτή, την υπερψήφισα, γιατί συμπεριλαμβάνει στρατηγικέ ενσωμάτωση και ένταξη για του Ρωμά. Στόχο μα είναι η στέγαση, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η απασχόληση για τι κοινότητε των Ρωμά. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθεσε ένα ακόμα ζήτημα, το ζήτημα τη μη εισαγωγή διακριτική μεταχείριση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρεθεί απαραίτητη χρηματοδότηση, θα πρέπει να προωθήσουμε προγράμματα και σχέδια τα οποία θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Ρωμά και παράλληλα όμω θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Άρα θα πρέπει να παρακολουθούμε του και τη χρήση των πόρων αυτών και να έχουμε και συγκεκριμένου δείκτε όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Πρέπει να πω ότι εκτιμώ όλου ιδιαίτερω τι προσπάθειε που καταβλήθηκαν προκειμένου να έχουμε και εκπροσώπου των Ρωμά στην όλη διαδικασία εκπόνηση τη έκθεση αυτή. Κυρίε και κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα πεπειραμένη στο ζήτημα της ενσωμάτωσης των Ρωμά στην χώρα μου, την Τσεχία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση των παιδιών των Ρωμά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στη γενικότερη ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον Άντζελ Ζαμπάσκη. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντω και εγώ ήμουν απεπισμένο ότι θα καταψήφιζα το ψήφισμα αυτό. Πρέπει να σταματήσει επιτέλου η υποκρισία που επιδεικνύουμε στον τομέα αυτό. Μιλάμε συνεχώ, γενικά και αόριστα, προτιμάζουμε ψηφίσματα και εκθέσει, αλλά δεν καταλήγουν σε τίποτα το σημαντικό, το ουσιαστικό. Τα γκέτο των Ρωμά εξακολουθούν και παραμένουν. Οι άνθρωποι είναι εκεί απομονωμένοι και δημιουργείται μεγάλη ένταση που σε βία, σε εγκληματικότητα, σε αποδόμηση των ίδιων των κοινωνιών εν τέλει. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε όλε αυτέ τι περιοχέ, όλα αυτά τα γκέτο. Στη δική μου τη χώρα, την Βουλγαρία, υπάρχουν και πάρα πολλέ επιθέσει κατά των αστυνομικών, κατά των ίδιων των ιατρών που πηγαίνουν στα γκέτο για να βοηθήσουν του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να εξαλειφθεί με ωραία ψηφίσματα ή γενικόλογε εκθέσει. Τα προβλήματα θα εξαφανιστούν μόνο όταν κατεδαφίσουμε τα αυθαίρετα κτίρια, όταν τα παιδιά αρχίζουν και πηγαίνουν στο σχολείο, όταν σταματήσουμε τα κοινωνικά επιδόματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο κατάχρησης από πολλούς Ρωμά. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Σα ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Σκρίπεκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη χαρά υποστήριξα το συγκεκριμένο ψήφισμα για την ένταξη του Ρωμά ε, σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας και σε όλους τους τομείς. Είναι ζωτική σημασία αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δούμε πώς συνεργάζονται οι διάφορες ομάδες στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο τα παιδιά και η παιδεία, αλλά και η ποιοτική στέγη. Ε, έχουν γίνει όμως πολλές επενδύσεις, έχουν αφιερωθεί πολλά κονδύλια σε αυτό το τομέα και εγώ πάντα απευθύνομαι στου εκπροσώπους στο Ρωμά και του καλώ να αξιοποιούν αυτέ τι καλές ευκαιρίε και να είναι σε επαφή με του θεσμού που στόχο έχουν να βελτιώνουν τι συνθήκε διαβίωση, στέγη, να δίνουν περισσότερε ε, ευκαιρίε στα παιδιά και να βελτιώνουν την κατάστασή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά ε, και να μην παραμένουν παθητικοί αποδέκτες ε, της βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα είναι αρκετά νυφάλαιο και δεν αναφέρεται πάρα πολύ ε, στην πλήρη συμμετοχή των ίδιων έτσι ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκρίπεκ. Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Σόσνιερτς. Ευχαριστώ. Σε αντίθεση με αυτά που διαβάζετε στην έκθεση, η Ρωμά ε, και η Τσιγκάνη, δεν υφίστανται ρατσιστικές επιθέσεις. Ο κόσμος τους αντιπαθεί, όχι επειδή είναι τσιγκάνοι, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο ζουν και φέρονται. Ο πολιτισμός τους, η κουλτούρα τους είναι πολύ διαφορετική πολλές φορές από την κουλτούρα των ε, μερών που ζουν. Και αυτό ε, είναι πολύ κακό επίσης να χρηματοδοτούμε τους Ρωμά επειδή είναι Ρωμά. Ε, τι προτείνετε δηλαδή εσείς ότι επειδή κάποιο έχει μια συγκεκριμένη καταγωγή ε, δικαιούται να εισπράττει και κονδύλια παρόλη την ε, ρητορική αυτή κατά των διακρίσεων, ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο κατά το Ρωμά, γιατί ρέουν τα κονδύλια και η αθρώα και δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Τα πράγματα μόνο χειρότερα γίνονται. Και αν ήθελαν, θα μπορούσαν να έχουν ενταχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στην κοινωνία, αλλά οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ζουν εκτός της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο τελευταίος ομιλητής για το θέμα αυτό, ο κύριος Πόλτσακ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή και είμαι πολύ ικανοποιημένο για το ότι εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμμερίζομαι την άποψη ότι ουδή θα πρέπει να αισθάνεται απομονωμένο, παραγωνισμένο στα πλαίσια τη κοινωνία. Κανεί δεν θα πρέπει να στερείται τι απαραίτητε ευκαιρίε για να οδηγηθεί σε προσωπική επιτυχία. Νομίζω ότι θα πρέπει σαφώ ρουσπαστικά να βελτιώσουμε τι δυνατότητε εκπαίδευση αλλά και απασχόληση των Ρωμά. Επίσης, η μη διάκριση θα πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε κοινότητα των Ρωμά οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα όμως, γνωρίζω ότι η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει και νέε προκλήσει. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε όλε τι στρατηγικέ μα προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τι απαραίτητε συνέργειε. Η κοινότητα των Ρωμά θα πρέπει βέβαια να γνωρίζει ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσει και θα πρέπει βέβαια και οι προσωποί τους να ενθαρρύνουν την αντίληψη αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, την έκθεση της κυρίας Ρουής, εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ζένελφετ έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, σύμφωνα με το άρθρο 9 για την συνθήκη και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 20, κάθε πολίτης της Ευρωπαϊ... ενός κράτους μέλους είναι και η πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, οι περισσότεροι στην Ευρώπη δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Δεν έχουν γνώση των δικαιωμάτων τους. Και αυτό το βλέπουμε αν αναλύσουμε τα ερευνητικά στοιχεία που δείχνουν ότι το 54% λένε ότι έχουν κάποια γνώση. Το 45% όμως των ε, πολιτών ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ιδέα ε, για το ποια είναι τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους, υποχρεώσεις τους, καθώς απορρέουν από την ευρωπαϊκή ηθαγένειά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλυφθούν δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Χρειαζόμαστε την ένταξη, την ασωμάτωση των Ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ζαμίτ Ευχαριστώ. Όταν ε, μιλούμε για την ηθαγένεια, πρόκειται για ηθαγένεια ω προ ένα κράτο μέλο, αλλά και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πολύ σωστά ε, η, έκθεση μιλάει και κάνει λόγο και για τα καθεστώτα πώληση διαβατηρίων. Όπω στην περίπτωση τη Μάλτα, λαμβάνει ένα μαλτέζικο ε, διαβατήριο, αυτό ισοδυναμεί με ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Από το 2014 αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται ε, τέτοιου είδους πώληση διαβατηρίων χωρίς να έχει κανείς ε, πραγματικούς δεσμούς με την χώρα που εκδίδει το διαβατήριο. Και πραγματικά είναι λυπηρό που κινείται με τέτοιο τρόπο η μαλτέζικη κυβέρνηση χωρίς διαφάνεια. Ξέρουμε ότι δύο οικογένειες από τη Σαουδική Αραβία αγόρασαν 62 διαβατήρια. Και τώρα η κυβέρνηση, καθώς πρόκειται και για θέμα ε, υπόλοιψης, ε, λένε ότι αυτά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για την κοινωνική στέγαση. Πρέπει όμως ε, να τηρούνται οι ευρωπαϊκές αξίες. Υπάρχει φυσικά και η αρχή της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ελέγξουμε αυτά τα καθεστώτα, αυτά τα προγράμματα, για να μην διακινδυνεύονται οι αξίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ας προχωρήσουμε στην έκθεση του κυρίου Λαμασού για την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία. Dear colleagues, we must be careful. Αγαπητοί συνάδελφοι, προσοχή με την ενισχυμένη συνεργασία. Πρώτον, ε, από την ίδια του τη φύση το εργαλείο αυτό υπονομεύει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επιπτώσεις εντός και εκτός. Δεύτερον, η ε, ομοφωνία ε, στο συνασπισμό των προθήμων σημαίνει ότι έστω και ένα κράτος μπορεί να διαφωνήσει και να βάλει ένα δούριο ύπο στη σχέση μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, είναι σχετική αποτελεσματικότητα. Κοιτάξτε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα έχει δικαιοδοσία στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτό. Η καταπολέμηση της απάτης λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι περιορισμένη, διότι οι χώρες αυτές ε, θα είναι ε, εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Υπερψήφισα την έκθεση, αλλά η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να στοχεύει στην πλήρη συνεργασία που είναι και ο απότερος στόχος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαμίκινς. Ε, και τώρα προχωρούμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Σπινέλη για την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για επεξήγηση ψήφου. Πρώτα κυρία Σόιτρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων αποτελεί μία από τι βασικέ αξίε που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα χάρτη που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ξεκάθαρα προ τα έξω ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα αποτελεί τη βασική αρχή για όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει πλήρη στήριση του χάρτη αυτού, χωρίς να υπάρχει καμία περιοριστική προϋπόθεση ως προς αυτό. Νομίζω όμως ότι ε, χρειαζόμαστε και ένα στρατηγικό κείμενο βάσει του οποίου υπάρχει και απαραίτητη προσαρμογή όλων των εσωτερικών κανόνων. Γιατί αν για παράδειγμα έχουμε εμεί ενδιάμεσε εκθέσει για το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τι δραστηριότητε εκπαίδευση και κατάρτιση ή για άλλε γραφειοκρατικέ διαδικασίε, τότε καταλαβαίνετε ότι ε, ο χάρτης αυτός χάνει την αξία του, δεν θα έχει καμία επιρροή στην ουσία. Γι' αυτό το λόγο απήχα κατά τη διάρκεια της ψηφορίας. Ευχαριστώ. Να μην Καλωσορίζω την έκθεση της συναδέλφου Σπινέλη. Πραγματικά στόχο ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι απλώ να αποφεύγουν ε, την ε, παραβίαση των συνθήκων, αλλά να διευρύνουν την εφαρμογή τη. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά που προτείνει η συγγήτρια είναι εκτός του χάρτη μελιωδών δικαιωμάτων. Συνεδριάσεις του Συμβουλίου ε, είναι κάτι το οποίο αποσκοπεί στο να μην βλέπουν οι πολίτες πώς παίρνουν οι αποφάσει. και χαίρομαι που αντέδρασε η διαμεσολαβήτρια. Δεύτερο, μιλάω για τους λεγόμενους τριμερεί διαλόγους αυτός ο όρος δεν αναφέρεται πουθενά στις συνθήκες και επίση ο κόσμος δεν ξέρει ότι είναι άτυπη αυτή η μορφή συνεργασίας. Ε, είμαστε προσιλωμένοι και εγώ προσωπικά και στη διαφάνεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και ε, γι' αυτό συμφωνώ να υπάρχει ξεχωριστή μελέτη αντικτύπου ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλη την νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Μαμίκινς. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση την έκθεση του κυρίου Ρανχέλ όσον αφορά το καθεστώ και τους γενικούς όρους άσκηση των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ο κύριο Ζένφελτ έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να θεσπίσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και μια σημαντική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εμείς επιλέγουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα γίνει Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Τα τελευταία όμως χρόνια, δυστυχώς, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό που είναι όμω ακόμα χειρότερο είναι ότι έχουμε εξάλληψη της ίδιας της δράσης συγκεκριμένων θεσμικών οργάνων, είναι και ίδιων των ίδιων των θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να προασπίσουμε σημαντικά θεσμικά όργανα στα κράτη-μέλη μας, όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν καταφέρνει πάντα να συνεργαστεί με τους συνηγόρους του πολίτη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτελούν ανάλογο έργο. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να στοχαστούμε πραγματικά αν θα πρέπει να έχουμε μια πιο συστημική, βιώσιμη λύση όσον αφορά την όλη επικράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Φόξ όσον αφορά μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Πολλοί ομιλητέ εδώ πέρα έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριο Μάιερ έχει πρώτο το λόγο. Κυρία. Η κυρία Μάιερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα με τα χαρά επισκέφθηκα ε, μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ε, μη επανδρομένα σκάφη ε, για να συλλέξει δεδομένα και μετά τα αναλύει. Η επιχείρηση έχει ήδη εντοπίσει πάνω από 20.000 ε, ε, ανομαλίες που ε, εντοπίζουν και ενισχύουν την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν τώρα νέες διαδικασίες που θα επιταχύνουν την ανάλυση και λένε κιόλα συγκεκριμένα ότι θα βγάλουν το ανθρώπινο στοιχείο από την εξίσωση. Βέβαια αυτό μπορεί να σημαίνει και την καταστροφή και απώλεια θέσεων εργασία. Εγώ πιστεύω ότι η χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μα βοηθήσει ε, αντιθέτω να δημιουργήσουμε περισσότερε νέε ε, νέες θέσεις απασχόλησης και νέε ευκαιρίε για ναι, τους εργαζομένους με δεξιότητε. Ευχαριστώ πολύ. μια σύνθετη βιομηχανική πολιτική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Είναι μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλία. Αυτό είναι και καλό και κακό. Αφενός είναι θετικό το ότι υπάρχει, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό ε, στις δραστηριότητε που απαιτούν μεγάλο όγκο γνώσεων και ε, δεξιοτήτων που έχει να κάνει και με το νομικό πλαίσιο που δεν ακολουθεί πλήρω ε, τι τεχνολογικέ εξελίξει. Ε, πολύ σωστά αναφέρονται στην έκθεση ζητήματα όπως ε, αυτά τη ευθύνη. Δεν πρέπει να τα υποτιμήσουμε. Υπάρχουν και ζητήματα δεοντολογίας που υπογραμμίζονται εδώ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των τομέων. Όμω, υπάρχουν σημαντικά κενά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την άμυνα και την ευθύνη για πολλές δραστηριότητες τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. και σε σχέση με μεμονωμένου πολίτε. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, ιδίω στον τομέα των νέων τεχνολογιών, γιατί εδώ έχουμε μείνει πολύ πίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε τέταρτο ε, των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στην ε, βιομηχανική δραστηριότητα και το ίμιση των ε, ρομπότ παροχής υπηρεσιών προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, αν εξετάσουμε τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή, την έρευνα ε, και ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νομοσύνη και τη ρομποτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε τόσο ε, καλοί σε αυτόν τον αγώνα. Η Κίνα και οι Πολιτείε προπορεύονται. Θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον του πολιτισμού μας. Και όχι μόνο στις υπηρεσίες ή στη βιομηχανία, αλλά και στην καθημερινότητά μας στην προσωπική μα ζωή. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη χάραξη πολιτικής και βιομηχανική πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό στηρίζω την έκθεση και θα ήθελα να υπάρχει μια πιο δυναμική προσέγγιση και ανάληψη δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Ταμπουράνο στην αίθουσα. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ. Στηρίζω την έκθεση του Ashley Fox για την ε, διασφάλιση μεγάλη πλειοψηφία σε αυτόν τον τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγάλε δυνατότητε ε, για την αύξηση τη αποδοτικότητα, ε, όμω υπάρχουν και προκλήσει. Γι' αυτό χαιρετίζω την έκθεση που λέει ότι απαιτείται ένα ε, σύστημα διαφάνεια και λογοδοσία σε ό,τι αφορά τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Ε, ενώ παράλληλα έχουμε και ω στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή ε, αυτή τη τεχνολογία και επιχειρήσει αλλά και πολίτε να εποφελούνται όσο γίνεται περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες πολλοί ευρωβουλευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και σε αυτό το φάκελο αλλά και σε άλλους έχουν τηρήσει μια συγκεκριμένη στάση και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Όμως ε, υπάρχουν ε, και ελλείψεις σε ό,τι αφορά το Brexit, οπότε καλό θα ήταν να το εξετάσουμε και αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος ομιλητή για την έκθεση αυτή είναι ο κύριο Σόσνιερτσε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή παραδέχεστε τελικά ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παράγουν το ίμιση των ιδιαίτερα εξειδικευμένων ρομπότ παγκοσμίω. Επομένω, αν τα πράγματα πάνε καλά, μην τα πειράζετε. Να σα υπενθυμίσω και μια έκθεση που είχαμε πριν από μερικού μήνε για την, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό εκείνων, ο οποίος ουσιαστικά επέφερε πολύ σημαντικές ζημιές όσον αφορά την ε, γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι και στην περίπτωση αυτή του γεωργικού τομέα και του βιομηχανικού τομέα στο παρελθόν είχαμε υπερρύθμιση, είχαμε υπερβάλλοντα αριθμό κανονισμών. Α μην κάνουμε το ίδιο σφάλμα και στον τομέα αυτό. Α μην δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλού κανονισμού οι οποίοι θα περιορίσουν τελικά την ε, ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να χάσει στον τομέα αυτό της τεχνικής νοημοσύνης εξαιτία τέτοιων κανονισμών. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Την έκθεση της κυρίας Γκούτελαντ όσον αφορά την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο Χαβιέρ Μπενίτο Τζελουάγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη ε, της Conservation, ε, θα μπορούσαν μετά από 100 χρόνια να έχουν εξαφανιστεί τα έντομα από τον πλανήτη. Τρομακτικό θα ήταν. Σήμερα το 1 τρίτο των ειδών εντόμων κινδυνεύουν με εξαφάνιση και θα ήταν ολέθριες οι συνέπειες αυτού του αφανισμού και για τα οικοσυστήματα αλλά και για την ίδια την ανθρωπότητα. Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν ότι η βασική αιτία του αφανισμού των εντόμων είναι σαφώς η χρήση φυτοφαρμάκων μαζί με τις εντατικές ε, πρακτικές ε, στις καλλιέργειες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει το γεωργικό μας μοντέλο με προληπτική προσέγγιση, να αποφεύγουμε την έκθεση σε ε, φυτοφάρμακα με βιώσιμες μορφές καλλιεργειών χωρίς χημικά, όπως είναι η αμυψισπορά, η φυσική και μηχανική έλεγχη, η χρήση φυσικών εχθρών. Απέναντι στη Μονσάντο θα πρέπει να έχουμε βιώσιμες λύσεις ε, ε, που θέλουν οι αγρότες και οι αγρότησες να υλοποιήσουν. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάθιος. ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία και ε, στην κυπουρική ε, και στην οποροκυπευτική είναι πάρα πολύ ε, απαραίτητη. Βεβαίως υπάρχουν και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα χημικά. Όταν ε, άρχισε ε, να κυκλοφορεί αυτή η ιδέα στο Κοινοβούλιο, εγώ την υποστήριζα. Αλλά ε, η έκθεση άλλαξε δρόμο και έχω αλλάξει κι εγώ γνώμη, γιατί ορισμένοι στόχοι και ορισμένα αριθμητικά στοιχεία είναι αβάσιμα. Πού είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Ακούμε διάφορα ουρανοκατέβατα που λανσάρουν ομάδες πίεσης και ομάδες συμφερόντων όπου θέλουν να ελέγχουν όλα τα χημικά που πηγαίνουν στη Γεωργία και ε, λέγουν ότι καταλήγουν ε, στον υδροφόρο ορίζοντα. Δυστυχώς αυτό είναι παράδειγμα κακής νομοθεσίας που τόσο συχνά χαρακτηρίζει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θα μπορούσε να είναι μια θαυμάσια νομοθεσία, δυστυχώς έχει καταλήξει έτσι ώστε να μην μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόιντροβα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή για τη βιώσιμη χρήση ε, των γεωργικών φαρμάκων. Συμφωνώ με τα κράτη-μέλη που ε, ότι πρέπει μάλλον τα κράτη-μέλη να διορθώσουν αμελητή τις αδυναμίες και τα προβλήματα που έχουν. Ε, Είμαι υπέρ των επενδύσεων στην έρευνα επίσης για να μπορέσουμε να βρούμε υποκατάστατα στα φυτοφάρμακα και καλύτερες εναλλακτικές ε, λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί ε, και η ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Τα γεωργικά φάρμακα ε, ε, ε, περιλαμβάνουν ουσίες και συστατικά που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να απαγορεύσουμε απολύτως και καθολικώς τη χρήση αυτών των χημικών. Και αυτό φορά και τις εισαγωγές από τρεις χώρες όπου έχουν καλλιεργηθεί τα προϊόντα με φυτοφαρμακά. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Σόλτες. Ευχαριστώ. Ε, σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη χρήση ε, των γεωργικών φαρμάκων και γενικά τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές συχνά στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως, ε, δεν διαφωνώ ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ε, στα τρόφιμα μπορεί να αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Όταν έχουμε κατάλοιπα στις ζωοτροφές, κάνει κακό στην υγεία των ζώων και πηγαίνουν και στην αλυσίδα των τροφίμων τελικά. Έχουμε δει πρόσφατα σκάνδαλα ε, τροφίμων. Ε, αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ε, υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Άρα θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο και χρήματα και ενέργεια και έρευνα στην ανακάλυψη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειας βιώσιμων, φυσικών, που καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας ήταν η βασική μορφή καλλιέργειας. Και επίσης θα πρέπει να είναι μικρές οι εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Το λόγο τώρα έχει ο, κύ... ο κύριος Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα όσον αφορά την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης. Η Γεωργία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα επίπεδο οικονομία υψηλό σε περιοχέ όπου δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική για την απασχόληση. Δυστυχώ όμω τα φυτοφάρμακα και εν γέννη τα γεωργικά φάρμακα έχουν έντονε περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορούν να αυξήσουν την σοδιά, αλλά μακροπρόθεσμα διαβρώνουν το έδαφο, καταστρέφουν κάποιου πολύ σημαντικού οργανισμού που βρίσκονται μέσα στο έδαφο και έχουν και άλλε αρνητικέ συνέπειε. Ήμουνα εισηγητή εκ μέρου των σοσιαλιστών όσον αφορά τη μελισσοκομεία και πρέπει να σα πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για τη χρήση τέτοιων χημικών ουσιών που επηρεάζουν έντομα όπω οι μέλισσε. Καλό λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου και να δώσουν προτεραιότητα στι επιλογέ τη μη χημικέ και τι μεθόδου εκείνε οι οποίε είναι λιγότερο επιζήμιε για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε σταθερά, βιώσιμα οικοσυστήματα, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση και για το ασφαλές περιβάλλον, αλλά και για τη βιώσιμη παροχή τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε έτσι στην, μάλλον στο τελευταίο μιλητή για την έκθεση αυτή, ο κύριος Μπόλτσικ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι η μακροπρόθεσμη μαζική χρήση φυτοφαρμάκων είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και για πολλούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάναμε το σημαντικό αυτό βήμα σήμερα. Η μαζική χρήση, όπως σας είπα, γεωργικών φαρμάκων έχει δραματικές επιζήμιες συνέπειες στο περιβάλλον. Διάβασα μια έκθεση πρόσφατα που λέει ότι πρώτο τέλος του αιώνα, μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα θα εξαφανιστούν όλα τα έντομα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό άμεσα συνδέεται με τη μαζική χρήση γεωργικών φαρμάκων και τα έντομα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα φάρμακα αυτά. Για να μην μιλήσουμε και την επίπτωση που έχουν τα γεωργικά φάρμακα στου ίδιου του ανθρώπου. Θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την έρευνα και την επιστήμη να βρούμε εναλλακτικέ μεθόδου λιγότερο επιζήμιε για το περιβάλλον. Να τονίσω επίσης ότι το περιβάλλον και δι' το βιώσιμο περιβάλλον θα πρέπει ως μέλημα να αντικατοπτρίζεται και σε όλες τι επιδοτήσεις που δίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία έκθεση είναι η έκθεση για την Μπελέτ μάλλον για ε, την ε, ολοκληρωμένη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η κυρία Κρούπα, σε ό,τι αφορά την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρέπει να πούμε ότι μπορεί να δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ε, σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες διασφάλισης της παροχής ε, υπηρεσιών υγείας στα κράτη-μέλη και διασυνοριακά. έχει να κάνει με την συμμόρφωση σε ό,τι αφορά την επεξεργασία πληροφοριών, ε, την περίθαλψη και τις υπηρεσίες που παρέχεται στους πολίτες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα γραφειοκρατίας, ε, ιδίω τα κρατημέλη πρέπει να τα αντιμετωπίσουν με τη δημιουργία contact points και για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την επιστροφή δαπανών. Η διασυνορική περίθαλψη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική ε, για όσους επάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Και η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι πολύ σημαντική στον τομέα ε, των διαγνώσεων και της ε, ιατρικής έρευνας. Και αναφέρουμε και την σημασία τη διασυνοριακή συνεργασία σε ό,τι περίθαλψη σε ό,τι αφορά τι πανδημίε και του εμβολιασμού. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριο Λενάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το δικαίωμα στη διασυνοριακή υπερίθαλψη είναι ένα από τα πλέον ε, σημαντικά επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα στι ε, μεθοριακέ περιοχέ, όπω το Λιμπούργο από όπου προέρχομαι. Ε, ε, μόνο να χάσουν έχουν οι πολίτε αν περιορίζει το δικαίωμά του στη διασυνοριακή περίθαλψη. Και αυτό δεν έχει δημιουργηθεί, ως, δεν έχει κατακτηθεί ω δικαίωμα από το πουθενά. Ε, και συνάδελφοι και που έχουν πάει μάλιστα μέχρι το Λουξεμβούργο στο δικαστήριο για να καταφέρουν ε, ε, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δαπανών τους. Όμω δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν την ταχύτερη δυνατή περίθαλψη όσο γίνεται πιο κοντά στο σπίτι τους, ακόμα και αν αυτό είναι στην άλλη πλευρά των συνόρων και θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, ε, για να άρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια ε, και να καταστήσουμε πραγματικά προσβάσιμη σε όλους τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λέναρς. Το λόγο έχει η κυρία Ρουχόνεν Λέρνερ. Κυρία Πρόεδρε, η ευμερία των ασθενών και το δικαίωμα στην ε, ποιοτική διασυνοριακή περίθαλψη ε, είναι κάτι το θετικό, γι' αυτό και είναι εύκολο να υπερψηφίσει κανεί μια τέτοια έκθεση, ε, γιατί υποφελούνται από αυτήν όσοι ταξιδεύουν σε άλλα κράτη-μέλη ή σε οποιονδήποτε άλλο που θέλει να υποφεληθεί τη περίθαλψη εκτό του κράτου μέλου του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τη δικασία επιπαραβάση κατά πολλών κρατομελών εξαιτία ε, παραλήψεων και ανεπαρκού εφαρμογή. Όλα τα κρατημέλη έχουν δηλώσει ότι έχουν υλοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτε να γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Το 2015 υπήρξε μια μελέτη που έδειξε ότι ούτε καν το 20% των Ευρωπαίων πολιτών ήξεραν και ε, είχαν επαρκή γνώση των δικαιωμάτων του ε, σε ό,τι αφορά ε, την υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την επίγνωση των δικαιωμάτων και μεταξύ των πολιτών και μεταξύ του ιατρικού προσωπικού. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο ομιλητή, ο κύριο Νέκοφ. Κύριε Πρόεδρε. Οι μεθοριακές ε, περιοχές καλύπτουν το 40% τη ευρωπαϊκή επικρατεία και πάνω από 30% των Ευρωπαϊκών πολιτών ζουν σε τέτοιες περιοχές. Ε, και στην Βουλγαρία έχουμε σύνορα με δύο με πέντε χώρε, δύο είναι ε, κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι μεθοριακέ περιοχέ δεν είναι πυκνοκατοικημένε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν υψηλέ ανάγκε ε, στην ιατροφαρμακευτική υπερήθαλψη, γιατί έχουμε και ένα γυράσκοντα πληθυσμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τι κατάλληλε υγειονομικέ δομέ. Βλέπουμε ότι τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια στην ε, Βουλγαρία, 19 μάλλον δομέ περίθαλψη έχουν κλείσει. Η διασυνορική περίθαλψη απαιτεί μια ειδική, απαιτούν, απαιτεί μια ειδική προσέγγιση και πόρους. Μία σημαντική πτυχή τη διασυνορική περίθαλψη είναι η έλευση ψηφιακών υπηρεσιών και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προ όλε τι αρχέ, ιδίω στι βουλγαρικέ, να υιοθετήσουν μέτρα για την εισαγωγή τη ε, ηλεκτρονική ε, υπαροχή υπηρεσιών των σύντομων δυνατών. Αυτό θα άρει γραφειοκρατικά εμπόδια και θα βελτιώσει την περίθαλψη σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε, κύριε Νέκοφ. Φτάνουμε στο τέλος ε, της ε, πρωινή ε, συνεδρίασης. Επιστρέφουμε στις 3.